Um Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας θα ήθελα. on the Εκεί πίσω στα ορεινά λίγη ησυχία. Λοιπόν, συμφωνούμε με την ημερήσια διάταξη. Ist man mit den Protokollen einverstanden? Με τα πρακτικά, επίσης. Ο συνήθως ανακοινός ο Πρόεδρος δεν έχει. Και πάμε μέσα στο σημείο 4 στην ημέρηση διάταξη. Απαλλαγή Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκήτρια έχει να κάνει τίποτα παρατηρήσεις. Αν όχι να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Ένα, σάκε, είπε. Τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο. είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ένα είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Die Abstimmung ist plus Ich habe has one extra. EFTD, ένας υπεράριθμος παρακαλώ να ρυθμιστεί. Λοιπόν, εγκρίνεται.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 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 51 ε, υπέρ 5, 7. Οι δύο που έχουν ξεχαστεί ε, και δεν έχουν την κάρτα τους είναι ο κύριος Γκάλερ και εγώ. Ερχόμαστε λοιπόν στην επόμενη έξι. Das ist jetzt der Menschenrechtsbericht, ne? Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Παντσέρη. Έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση πριν από την ψηφοφορία. Προτού αποφασίσουμε για την έκθεση. Όχι, εντάξει. Ξεκινάμε. Λίγη ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα. Ο κύριος Λίτς επίσης συμπεριλαμβάνεται στη σύσταση αυτή. Εξετατέσσερα ψήφι υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παρακαλώ. Χωρίς... Όχι, come on, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε είπαμε. 70 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα που χωρίς τις λέξεις among the member states and ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα για τις λέξεις αυτές. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 80 σε τμήμα, σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα ψήφι χωρίς λοιπόν τις λέξεις που έχουν προσθεθεί κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα φυσικά και απορρίπτεται και αυτό το δεύτερο τμήμα. 81 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 83 σε δύο τμήματα. Με τις, χωρίς τις λέξεις specifically among the Middle Eastern countries, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα για τις λέξεις αυτές με τις λέξεις αυτές υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία Ε, δύο υπεράριθμοι στους σοσιαλιστές. Κύριε είναι επιβάλλεται κάποια τάξη, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. «24 υπέρ 37 κατά και μία αποχή απορρίπτεται». «84 πάλι σε δύο τμήματα». Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Πιστεύω ότι είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Απολύτεται. 85 και 86 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές δεκτές. 87 υπέρ, κατά αποχές. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 σε δύο τμήματα. <clears throat> Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά έλεγχος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 91 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 93 <clears throat> υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχέ έλεγχος. Abstimmung 25 με 35 και 2 αποχές. 26 μάλλον. Απορρίπτεται. Ούτως ή άλλως. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ο 98 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 104 υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θέλουμε έλεγχο στην 104.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 κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται ε, εκπίπτει 116 συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές κάνουμε ελέγχο Πέρας ψηφοφορίας 34-35 34-35-128 28 με μία αποχή εγκρίνεται Εγκρίνεται. Πού ήμασταν τώρα. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παντσέρι 130. Μία χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος βεβαίως.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 κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. 33 με 30 και μία αποχή εγκρίνεται. 134 ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 136 πέρα κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ 170 είχε πει ο στην αρχή 140 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστή 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 31 zu 22. 31 με 22 δεκτή. 160 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160. 160. Αποχές δεκτή. 162 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά έλεγχος Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 34 με 26 και 3 αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρώτη σειρά των σοσιαλιστών έχει μια εντυπωσιακή συμπεριφορά 170 ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές ανεδεκτή. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 ναι 177 έλεγχος Abstimmung Απορρίπτεται. 31 υπέρ, 32 κατά και 3 αποχές. Απορρίπτεται. Κοιτάξτε, 31 υπέρ, είπαμε 32 κατά, έχει απορριφθεί. Δεν έχει την κάρτα του μαζί του ο κύριος Γκάλε. Εξάλλου και με ισοψηφία απορρίπτεται. 179 υπέρ. Α, 178 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Άποχες. Το αυτό. Έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται 32 υπέρ 30 κατά. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε. 182. 34 υπέρ, 30 κατά μία αποχή εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. 185 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10, όχι, όχι, όχι. Μια στιγμή, έχουμε και άλλη σελίδα. 191 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά έλεγχος 196 έλεγχος Abstimmung 30 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 198. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 24 υπέρ, 30, 25 υπέρ, συγγνώμη, 37 κατά απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 2.13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα μια στιγμή 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.23 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ. Ελέγχουμε. 223. Παρακαλώ. Κατά. τις geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. 35 υπέρ, 25 κατά. 2,24 υπέρ κατά αποχές Απόρριφτεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 226 πέρα Απορρίπτεται. 27. Χένκελ. Υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέ. κατά αποχές εγκρίνεται 232 υπέ. κατά έλεγχος για τη 232 Abschluss. Jetzt geschlossen. 34 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 239 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ. Κατά. Withdrawn λέει. Α, έχει αποσυρθεί καλά. 241 τότε. 241. Υπέρ. Κατά. Αποχές Τσεκ. Καλό. Πέρασε. Δεν κρυθηκε 34 34-27. 243, πέρα. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Closed. Mit 34 30. εγκρίθηκε. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 246 υπέρ. Βίσκι. Αυσίγουρες κυφλός. Ναι, ναι, ναι, ναι. have people left? Not one. Nobody has left. Seven people have not yet voted. Επτά δεν έχουν ψηφίσει. So, closed. Abgelehnt mit 30 zu 30. Απορρίπτεται ισοψηφία 30-30. Όχι 30-31. Εν πάση περιπτώσει και με ισοψηφία απορρίπτεται. 247 υπέρ κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Πρώτα ψηφίσουμε τη 246. Μα τη ψηφίσαμε τη 246. Load again. Someone is confused, nobody knows who. Δεν ξέρω, κάποια σύγχυση επικρατεί. 2.46. 2.46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 2.47 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 2.42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. Ist mit Πέρας. 35 υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. 2,48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας. 34 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται. Και ερχόμαστε τώρα στις 2.51 τροπολογία στην επόμενη σελίδα 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 259 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 260 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ υπέρ κατά αποχές έλεγχος Πέρας. 27-35 απορρίπτεται. 2-64. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2-65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2-66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2-67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2-68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ κατά αποχές 271 υπέρ και πάλι κατά και πάλι Πού να ξέρω. Έλεγχος. Abstimmung ist geschlossen. ψηφοφορίας. 33-32 εγκρίνεται. 2,72 υπέρ. Κατά αποχές. 2,73 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2,74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 276 υπέρ κατά αποχές απολύτωται 277 κατά αποχές απολύτω. 280 υπέρ κατά αποχές απολύτω. 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 279 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.81 2.82 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές έλεγχος Geschlossen. Πέρασε ψηφοφορία. 31-30. Εγκρίνεται. 283 dafür. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 284. 284. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 329, 29 εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ερχόμαστε στην 286 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 287 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 288 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 289 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς τη λέξη especially και μετά με τη λέξη especial. Με το χωρίς especial, με δίχως especially. Ψήφι Τώρα το especially, το ιδίως. Ψήφι Το ΕΛΚ ε, υποστηρίζει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα, βεβαίω. Especially. Das war doch klar abgelehnt, Πέρασε. 23 με 33 απορρίφεται 2,91 υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές απορρίφεται 2,90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 296 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Δύο λέει ο πρόεδρος. Πέρασε ψηφοφορίες. 36-28 εγκρίνεται. 2,97. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 304 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται συγγνώμη 306 υπέρ κατά αποχές δεκτή 307 υπέρ κατά αποχές δεκτή 308 υπέρ κατά αποχές δεκτή 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Όχι. Για το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Και πάλι. Κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. 30 με 33 απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 312 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 313 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 314 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για 315 πυρίζος. Η Abstimmung ist geschlossen. Πέρα. 31 <clears throat> με 33 απορρίπτεται. Ich doch gesehen. 316. <laughs> 316. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 323 υπέρ κατά αποχές δεκτή 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 υπέρ κατά αποχές δεκτή η πρώτη σειρά των σοσιαλιστών δεν ψηφίσει πια 326 υπέρ 326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 330 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3.31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.66 λέει ο, ο πρόεδρος 3.33 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3.34 είναι γλωσσική. 3.35 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3.36, 37 αλλά και 38 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά αποχέ έλεγχος. Ένα υπεράριθμος στο, στο ΕΡΤ, κύριε Γκάλερ. Πέρας ψηφοφορίας. 28 με 36 απορρίπτονται οι τρεις αυτές τροπολογίες. 3.39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 3.40 και 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 3.42 υπέρ. Κατά αποχές 3.42 επαναλαμβάνω υπέρ 3.42 κατά κανείς ηλεκτρονική επαλήθευση Abstimmung geschlossen. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει. Ας μην, ας μην σταθούμε στο προηγούμενο θέμα. 3.43. Πέρας. 343. 3.43, υπέρ. Κατά. Λοιπόν, ηλεκτρονικά. 343. 343 ηλεκτρονικά. Πέρας. 11 με 49 απορρίπτεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. 3.49 31 με 33 απορρίπτεται 350 υπέρ κατά αποχές δεκτή 351 υπέρ κατά αποχές δεκτή 352 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές δεκτή 354 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 357 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 355 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 356 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 358 υπέρ. Δεν χρειάζεται να την ε, ψηφίσουμε γιατί έχει εγκριθεί.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 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 368 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 369 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 370 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 68 3, 71, 72, 73, 74, 75 και 90, ποιο είναι το θέμα εδώ, ρωτάει δηλαδή, τη γραμματεία ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Αλλιώ Τζον Μπάσκι, Γκριλ, Μπλε, Χέγκελ, Σομπράτ και Μικολάσιτ Υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτώνται 378 υπέρ. Κατά. Υπέρ μάλλον. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ έχει ρυθμιστεί 381 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 383, 84, 85 και 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 387 υπέρ κατά απορρίπτεται 388 υπέρ κατά απορρίπτεται 389 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.90 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 390 για την 390 πέρας 35 με 29 εγκρίνεται 391 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σύμβαση 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 397 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 404 υπέρ κατά αποχές αυτό θέλει ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι ψηφίζετε. Πέρας. Είκοσι 34 ε, κατά, απορρίπτεται. 21 υπέρ, αλλά δεν έχει σημασία. 405 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 20 κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Τσεκ, ελέγχουμε. 413. Check is Πέρασε το ελέγχο. 33 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται. Πού είμαστε τώρα, τις 4.13 έτσι. 4.14 υπερ Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται νομίζω. 4.15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται, 4-16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται, 4-17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 18 dafür. 418 υπέρ. Dagegen Enthaltung angenommen. Κατά αποχές εγκρίνεται. 419 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 421 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Λοιπόν, πού πού τώρα, 423. Πάμε 424 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αν νομίζω ότι είχε απορριφθεί. Abstimmung Πέρας. 32 υπέρ 33 ε, κατά απορρίψεται. 425 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.28 υπέρ όχι την καταπέμπτει, όχι την ψηφίζουμε 4.28 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 427 ειπε Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 430 υπέρ. Κατά αποχε εγκρίνεται. 433 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 436 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 432 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 417 υπέρ 17, όχι, συγγνώμη, 4.37 διορθώνει ο πρόεδρος, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, όχι, εγκρίνεται. 4.35 είναι γλωσσική, 4.38 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4.39 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Δηλαδή εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Έλεγχος, καλά. 4.39. Abgeschlossen. Πέρασε. 32 υπέρ, 31 κατά εγκρίνεται. Ε, 441 γιατί καταπίπτει προηγουμένη. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 442 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4, 43 όχι, 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 445 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 446 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 447 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία υπαρίθμα 450 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 451 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 452 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Abstimmung ist geschlossen. Peres. Mit 32 zu 29. 32 υπέρ 29 κατά εγκρίνεται. Οι επόμενες υπέρ 453, 54, 55 κατά αποχές απορρίπτονται. 456 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Έχουμε μια προφορική εδώ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 457 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 459 υπέρ κατά αποχές ξανά 459 παρακαλώ ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές ενέ 460 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 462 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 464 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 466 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρασε. ist geschlossen. Mit, was war das jetzt? Τι έχουμε τώρα εδώ. 32-32 ισοψηφία απορρίπτεται. 467. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 469 υπέρ. Υπέρ. 469. Κατά. Εγκρίνεται. 470 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 74, ε. Πέρας. 28 υπέρ, 32 κατά, 471 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 472 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 473 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 474 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 475 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 476 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 477 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 478 υπέρ 477 έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικά. 29 υπέρ 36 κατά αποχές. Κυρία Λόχ Μπίλερ, να με πιστεύετε λίγο παραπάνω, παρακαλώ. 4,78 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. 4,79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. 85 λέει πάμε τώρα και πού είναι αυτή να τη βρω. Όχι, λάθος. Στην 486 πάμε, λέει ο πρόεδρος. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εδώ χρειάζεται παλήθευση. Ό,τι να είναι είναι. Das 43, ne? 30 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 46 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 είπε κατά Αποχές έλεγχος παρακαλώ για τη 48. 29 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίψεται 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίψεται 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίψεται 56 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 είναι γλωσσική στο περιεχόμενο Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε ίσως κάποιες τροπολογίες. Θέλετε τσεκ. Τι να κάνω, ούτε η ίδια μου η ομάδα δεν με πιστεύει. Του glaubst mir <laughs> Πέρα στην ψηφοφορία για την 63. 33-27. 33-28 εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά απορρίπτεται. Τρία υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά χες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 Μπορούμε να ψηφίσουμε τις πρώτες τέσσερις μαζί. ΔΒ1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. ΔΒ2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΒ3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΒ4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά έλεγχος. ΔΕΒ 7. Χωρίς μικρόφωνο πέρα της ψηφοφορίας 33 με 27 δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ 20 θέλετε έλεγχο βεβαίως ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας ναι ναι είναι φανερό δεν, δεν έγινε δεκτή 11.49 απορρίφθηκε 20 11.50 πράγματι 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Επιτροπή Γυναικών 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τι είναι 21 τώρα ωραία Εξέπεσε 2, πάμε στην 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θεέ μου λέει ο πρόεδρος δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο Μπορούμε να ψηφίσουμε από την 5 έως τις 16 από κοινού. Ναι. Ναι ή όχι. 5 με 13. Εντάξει. Ψήφι υπέρ. 5 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται 6 υπέρ κατά απορρίπτεται 7 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται 8 υπέρ κατά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 κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται 20 υπέρ κατά αποχές για την 20 επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος για την 21. Πέρας. 34-28 δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά από 24 υπέρ κατά από απορρίπτεται 25 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ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 αποχές 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ 51 έλεγχος. Πέρας. 34 με 27 δεκτή. Αυτή ήταν η 51. 52. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 54. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε την τελική ψηφοφορία. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι σωστό όταν μια επιτροπή που είναι γνωμοδοτική προσπαθεί να ξαναγράψει όλη την έκθεση. 55 τροπολογίες δεν νομίζω ότι αυτό έχει νόημα. ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία λοιπόν άρχεται. Πέρας. 49 υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. E η ομαδα ecr εχει να καταθέσει ε, μια ψήφο, μια ψήφο μειοψηφίας. Πρέπει να το πω από την αρχή. Έχουν στείλει επιστολή κάποιοι συνάδελφοι αν θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Εξαγγέλθηκε την περασμένη φορά και δεν διαφώνησε κανείς. Οπότε και θα προχωρήσουμε στη συζήτηση όπως προβλέπει η ημερησία διάταξη.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 name, Σας παρακαλώ καθίστε. Οι συνάδελφοι που θέλουν να αποχωρήσουν ή οι επισκέπτες παρακαλούνται να αποχωρήσουν σε αιθούσεις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 Hmm? 15 minutes is fine? Dear colleagues, meine Damen und Herren. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες μου και κύριοι, καλωσορίζω ε, νόπιον μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της ε, Ρωσικής Κρατικής Δούμα, τον κύριο Αλεξέη Πουσκόφ. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν και η παρούσα συνεδρίαση συνέχιση προηγούμενης συζήτησης. Θα μιλήσει ένα τέταρτο ο ίδιος και μετά έχουμε τρία τέταρτα για τη συζήτηση στη διάθεσή μας. Σημειώνω ε, ε, όσους θέλουν να μιλήσουν και αναλόγως με τον αριθμό θα μοιράσουμε και το χρόνο ομιλίας για να μπορέσετε να μιλήσετε όλοι. Ξέρουμε ότι γίνεται αυτή η συζήτηση σε καιρούς που είναι τα πράγματα πάρα πολύ τεταμένα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συμμετείχα στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, όπως και μερικοί από εσά και διαπιστώσαμε ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά αποφασιστικής σημασίας. Όταν ε, σας καλέσαμε δεν ξέραμε ότι θα ζούσαμε τόσο συναρπαστικούς καιρούς. Δεν έχετε διερμηνία. Ε, Wir Γνωρίζουμε ότι οι εντάσεις αυτές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ε, ελπίσουμε ε, στα πλαίσια της Συμφωνίας της Νορμανδίας να βρεθεί μια φόρμουλα να γίνει συνάντηση στο Μίνσκ. Ορισμένοι λέγουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για να φτάσουμε σε ειρηνική λύση πριν αρχίσουν κάποιοι να ε, δίνουν όπλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σαφή ε, πλειοψηφία σε ένα ψήφισμα έχει ε, λάβει θέση και εμείς θέλουμε να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την προσάρτηση της Κρυμαίας και στη συμμετοχή της Ρωσίας ε, στην Ανατολική Ουκρανία θεωρούμε ότι είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο, ε, οι ε, κυρώσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και να επιβάλλονται όσο δεν τηρεί τη συμφωνία του Μίνσκ και δεν εφαρμόζεται και η υποστήριξη των ε, Ρώσων προς τους αυτονομιστές και η ρωσική ανάμιξη όπως τη βλέπουμε εμείς. Βέβαια ο κύριος Πουσκόφ θα διαφωνήσει θα πρέπει, ε, ε, θεωρούμε ότι όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι παραβίαση και κόλαφος για τη Συμφωνία του Μίνσκ. Ε, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα είναι πάγια θέση μας αυτή, ενδιαφέρεται για να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία και είμαστε πάντα πρόθυμοι να άρουμε τις κυρώσεις και να αρχίσει να επαναληφθούν οι ε, συζητήσεις για την Συμφωνία Εταιρική Σχέσης, για τον εξχωρισμό της ρωσικής οικονομίας και μερικά άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να τα λέμε δημόσια, αλλά υπάρχουν και όροι και προϋποθέσεις να επανέλθει το διεθνές δίκαιο εκεί και θεωρούμε ότι με τη Συμφωνία του Ελσίνκη, την πράξη, τη χάρτη του Παρισίου, ε, το μνημόνιο της Βουδαπέστης και μερικά άλλα πράγματα που φέρουν τη ρωσική υπογραφή εξασφαλίζεται και θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να επανέλθει η εδαφική ακαιρεότητα και ιδιαίτερα το θέμα που έχει να κάνει με τα ε, κυριαρχικά δικαιώματα κάθε κράτους να αποφασίζει ελεύθερα με ποιον συνάπτει συμβάσεις και συνθήκες. Και δεν υπάρχουν θέματα της εγγυη αλληλοδαπής και τέτοια. Τι να. Αλεξέη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για μια επιχειρηματολογία με τρία σημεία ότι έχουμε ιστορικές εκεί αξιώσεις ή ε, τα συμφέροντά μας ασφαλείας δεν διασφαλίζονται ή ε, ε, παραβιάζονται υποφέρουν διάφορα δυνάμει ονότητε, πράγμα που δεν ισχύει στην Ουκρανία γιατί υπάρχει και το Συμβούλιο της Ευρώπης γι' αυτό. Ε, με τέτοια επιχειρήματα ε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να αναφλεγούν. Και είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν θα γυρίσουμε στην καμαρίλα ε, παρελθόντων των αιώνων και σε τέτοιες πολιτικές που οδηγούσαν σε πολέμους. Βεβαίως είναι θέμα της κυριαρχίας αυτό, της ελεύθερης βούλησης όχι μόνο του Ουκρανικού λαού αλλά ε, είναι και ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και θα πρέπει να επανέλθει η ομαλότητα εκεί γιατί στο και το αντίθετο θα οδηγεί στην Ευρώπη σε ανασφάλεια και σε ε, καταστάσεις επικίνδυνες που θεωρούσαμε ότι είχαμε ξεπεράσει τα τελευταία 25 χρόνια. Και όταν έχεις λανθασμένη άποψη για τον αντίπαλο ή θεωρείς ότι δεν φέρεται σωστά, δεν είναι ε, δικαιολογία για να παραβιάζεις την εδαφική του ακαιρεότητα. Οπότε είναι παράδεκτο για μας αυτό. Νομίζω περιέγραψα πώς βλέπουμε εμείς την κατάσταση με τρόπο σύντομο ευσύνοπτο και νυφάλιο και ελπίζω να ε, έχουμε τώρα τη δυνατότητα με βάση αυτά να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση και θα πρέπει να λάβουμε και τις ευθύνες μας απέναντι στους λαούς από τους οποίους έχουμε εκλεγεί. Αλεξέη, έχεις το λόγο. Thank you, Elmer. Thank you, Elmer. Ευχαριστώ, Elmer. δέχτηκα την πρόσκληση του κυρίου Μπροκ. Γνωριζόμαστε εδώ και καιρό. Γνωρίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια πλειοψηφία που δεν έχει ακόμη διατυπώσει μια τελική θέση. Και φανταζόμαι ότι δεν είναι και το πιο εύκολο κρατήριο αυτό στο οποίο απευθύνομαι. Μια εύκολη λύση θα ήταν να μην έρθω και να μην δεκτώ κάποια κριτική ή κάποιες επιθέσεις που σίγουρα να μένω. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι αν και είναι έντονα τα συναισθήματα και φυσικά αυτή τη στιγμή οι κατηγορίες ε, δημιουργούν πολιτική. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε εκ του μηδανός. Θέλω να υπογραμμίσω την ετοιμότητα του κ. Λέντ και της κ. Μερκέλ να αναλάβουν μια νέα πρωτοβουλία ενώπιον μιας κατάστασης που μπορεί να φύγει εντελώς εκτό ελέγχου και γι' αυτό ήρθα στο Στρασβούργο. Και γι' αυτό τώρα απευθύνομαι εδώ σε εσά, όχι για να μπω σε έναν ιδεολογικό πόλεμο εναντίον σα, δεν είναι ο στόχο μου αυτός, ούτε να σα κάνω να δεκτείτε τη ρωσική σκοπιά, δεν είναι ο στόχο μου αυτό. Υπάρχει μια παροιμία γαλλική ότι πρέπει να ε, ε, πείσουμε τους πεπισμένους. Είναι δύσκολο να πείσουμε κάποιους που πιστεύουν κάτι διαφορετικό. Και ήθελα να σας αναφέρω κάποια στοιχεία της κατάστασης, ε, τα οποία χρειάζονται μια νέα προσέγγιση και δεν είναι, εδώ να προβούμε σε αμοιβές κατηγορίες, γιατί αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Καταρχήν ε, πιστεύω ότι η συνάντηση στο Κίεβο και στη Μόσκα, οι συναντήσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικές γιατί ο πόλεμος αυτός δεν πηγαίνει πουθενά. Είναι ένας πόλεμος που θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ καιρό ε, σε χαμηλή ένταση, όπως έχει γίνει από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου ε, με κάποια κρούσματα έντονη σύραξη. Όμως θα μπορούσε να είναι και ένας πολέμος που θα διευρυνόταν και θα αποτελούσε πράγματι μεγάλο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μάλιστα εξετάζουν τη δυνατότητα να στείλουν όπλα στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια εξέλιξη επικίνδυνη και θα συμφωνήσω με τον Λαντ που είπε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολικό πόλεμο. Επίση ξέρουμε πώ ξεκινούν αυτά τα πράγματα. Καταρχήν φτάνουν τα όπλα, κατόπιν στρατιωτικοί σύμβουλοι. Στη συνέχεια έχουμε στρατεύματα για να του υπερασπίσουν. Κατόπιν έχουμε ανθρώπου που σκοτώνονται και έχουμε ε, μια πλήρη στρατιωτική εμπλοκή. Όπως ξέρουμε από την ιστορία του Βιετνάμ, έτσι ξεκινήσε ο πόλεμος του Βιετνάμ με την αποστολή όπλων και κατόπιν είχαμε ένα πλήρη πόλεμο. Είναι πολύ επικίνδυνη λοιπόν η κατάσταση και δεν πιστεύω ότι διαφορετικά ο καγγελέρος της Γερμανίας και ο πρόεδρος ε, της Γαλλίας ε, θα είχαν ε, αρχίσει να εργάζονται επί της, της πρωτοβουλίας με μια τόσο σοβαρή προσέγγιση όπως έχουν σήμερα. Το να σταματήσουν τώρα οι είναι κρίσιμο, είναι ζωτικό. Και ο λόγος είναι γιατί ε, πολλοί άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε εχθροπραξίες πεθαίνουν στην Ουκρανία. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται από τους αντάρτες λέγεται, όμως αυτό σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αλήθεια. Παραδείγματο χάρη, θα σας δώσω τα νούμερα για την τελευταία εβδομάδα στον Τόνεσκ. 105 κτίρια, κατοικίες καταστράφηκαν, 3 νοσοκομεία, 2 σχολεία, 2 νηπιαγωγεία, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και 100 τραυματίστηκαν περίπου. Σίγουρα αυτό δεν γίνεται από τους αντάρτες γιατί αυτοί ελέγχουν τον Τόνες και γιατί να το κάνουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μια ανταλλαγή. Φυσικά η Ουκρανική πλευρά θα δώσει τα δικά τη αριθμητικά στοιχεία. Και δεν λέω ότι σε αυτό το πόλεμο υπάρχουν καλοί και κακοί. Λέω ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμο αυτό, γιατί τα επίσημα νούμερα είναι ότι 5.300 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους και 10.000 έχουν τραυματιστεί. Αυτά είναι νούμερα του ΟΗΕ. Οι μυστικές υπηρεσίες της ε, Γερμανίας έχουν δώσει κάποια άλλα νούμερα ε, ότι 50.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία και αυτό θα πρέπει να μας ε, κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Πού πάμε από εδώ και πέρα, θα πολυπλασιάσουμε τα νούμερα αυτά ή θα πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς ότι σε αυτό το πόλεμο αν δεν υπάρχει μια διεθνής πολιτική επέμβαση μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Όπως ξέρετε, όλοι οι πόλεμοι δημιουργούν και στις δύο πλευρές ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν μέχρι το τέλος, ρίζος πάστες. Θα το βρείτε και στο Κύβολα και μεταξύ των εντερτών. Πάντα συμβαίνει αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι που ακούγονται πολύ πεπισμένοι, αισθάνονται ότι έχουν δίκιο. Αναρωτιέμαι όμως, στην περίπτωση της Ουκρανίας, πού είναι Πού θα τελειώσει αυτό, θα μπορέσουν να πάρουν το κύβο, οι εντάρτες δεν θα μπορέσουν να πάρουν το Κύβο, αυτό είναι προφανές και δεν έχουν και το στόχο αυτό. Όμως αν πολεμήσουν ε, μέχρι τέλους ε, οι Ουκρανοί, τι θα κάνουν τελικά, θα σκοτώσουν όλους τους αντάρτες. Δεν νομίζω ότι και αυτό μπορεί να γίνει. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αλλά και τον Ιανουάριο είχαμε επιθέσεις από το Κίεβο και ε, από τώρα έχουμε ένα status quo στον πόλεμο αυτό. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Καμία πλευρά δεν ε, μπορεί να ζημιώσει αποφασιστικά την άλλη πλευρά. Επίσης ήταν πολύ απλό να πούμε ότι είναι η κατάσταση άσπρη και μαύρη. Δηλαδή είναι μαύροι οι αντάρτες, είναι οι κακοί και οι καλοί είναι στο Κίεβο. Στην τελευταία εβδομάδα υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα από το Κίβο που ε, αποκάλεσε τη Ρωσία ως ε, μια χώρα που εξαπολύει επίθεση στην Ουκρανία. Η ερώτηση μου είναι... Έχετε δει πολλές επιθετικές χώρες ε, που θα δέχονταν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην επικρατεία τη Αν η Ρωσία επιτίθεται γιατί χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν Καταφυγείο στην ρωσική επικράτεια, αν πρέπει από την Ουκρανία. Δηλαδή αυτό δεν εντάσσεται σε αυτήν την ασπρόμαυρη εικόνα και να σα πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι είναι κυρίω Ρώσοι και αισθάνονται πιο ασφαλεί σε ρωσικό έδαφο. Ταυτόχρονα περίπου 120.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές ε, και έχουν βρει καταφύγιο σε άλλες περιοχές στην Ουκρανία. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και ένα χάσμα στην Ανατολική Ουκρανία. Κάποιοι θα προτιμούσαν να πάνε στη ρωσική πλευρά και κάποιοι στην Ουκρανική πλευρά. Και ακριβώ επειδή δεν είναι άσπρο και μαύρη εικόνα, χρειάζεται πολιτική λύση. Και ακριβώ επειδή ζουν εκεί στην Ανατολική Ουκρανία περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πιστεύουν και αυτοί. Γι' αυτό η ερώτηση του μελλοντικού ε, στάτους, ε, του καθεστώτος ε, αυτής της επικράτειας είναι κάτι θεμελιώδες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η μοίρα του θα αποφασιστεί μόνο στο Κίεβο. Φοβάμαι ότι η Ουκρανική κρίση έχει γίνει διεθνής κρίση. Δεν υπάρχει μόνο μια εγχώρια λύση, έχει γίνει μεγαλύτερη από αυτό δυστυχώς. Και Νομίζω ότι το θέμα του καθεστώτος, του στάτους είναι η βάση επί την οποία μπορούμε να έχουμε όχι απλώς μια εκεχηρία που θα παραβιαστεί σε μία ή δύο εβδομάδες, αλλά να έχουμε μια διαρκή ειρήνη. Γιατί οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα πρέπει και αυτοί να πουν τη γνώμη τους, να τοποθετηθούν για το ποιο καθεστώς θα θεωρήσουν ότι εγγυάται τα δικαιώματά τους και τις προσδοκίες τους. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς χωρίς να τους ρωτήσουμε. Και δεν ακόμα από το Κίεβο. Το ίδιο μότο θα λέγαμε, θα μείνει μια νέα χώρα η Ουκρανία. Ναι, είναι το δικαίωμά τους να το λένε αυτό, αλλά θα δούμε και την κατάσταση. Μια νέα χώρα ε, μπορεί πάντοτε να ανταποκριθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικέ κοινωνίε στη Σερβία στην ε, εποχή τη κρίση με το Κουσουπέδιο. Είχαμε κάποιου ζουσπάστε που έλεγαν ότι θα πρέπει να μείνει ενωμένη η Σερβία. Να μείνει ενιαία. Μα οδήγησε αυτό. σω αν είχαμε ένα ομοσπονδιακό καθεστώ για το κοσμοπέδιο θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα και ίσω είχαμε πολύ λιγότερα θύματα στη Ιουκοσλαβία. Δεν προτείνω λοιπόν η Ουκρανία να γίνει απαραίτητο μια ομοσπονδία και δεν βλέπω κανένα πρόβλημα με την ομοσπονδία όπως και πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί. Η Γερμανία είναι ομοσπονδία, η Ρωσία είναι ομοσπονδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ομοσπονδία. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι κακό με αυτό. Όμως εγώ σίγουρα θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώ για την περιοχή αυτή που θα γίνει αποδεκτό από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί. Δεν θα αποφασιστεί αυτό στην Ουάσιγκτον, στη Μόσχα, στι Βρυξέλλε ή στο Κίεβο. Πρέπει να ρωτήσουμε του ανθρώπου αυτού και θα πρέπει αυτοί να τοποθετηθούν και να πούν ε, ποιο καθεστώ θα ήθελαν. Για τον Ντόν Μπάς, ναι, θα πρέπει να μείνει μέρος της Ουκρανίας. Δεν ε, διαφωνούμε με αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, από όλες αυτές τις καταστροφές και τους θανάτους και τις σκληρές χειροπραξίες, δεν πιστεύουμε ότι απλώς μπορούμε να πούμε στο Κίεβο εντάξει, θα έχεις ένα νέο κράτος, κάνω ό,τι θέλεις εκεί, θα υπάρχουν εκδικητικές πράξεις, θα υπάρχουν παράνομες ε, πράξεις κατά των κατοίκων και θα πρέπει να τους δώσουμε κάποιες εγγύσεις ασφάλειας για τις εγγύσεις αυτές πιστεύω ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπαθειές μας. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του Κιέβου έχει δημιουργήσει σχετικά στενούς δεσμούς με αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν παραδείγματο χάρη η κατάπαυση του πυρός από την πλευρά του Κιέβου την εγγυηθούν την κατάπαυση ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια απάντηση φυσικά από την πλευρά μας. Η Ρωσία θα μπορούσε να ασκήσει μια επιρροή στους αντάρτες έτσι ώστε να διαρκέσει αυτή η κατάπαυση του πυρός και να μην παραβιαστεί πολύ σύντομα. Και επίσης αυτές οι εγγυήσεις που πιστεύω ότι θα εξεταστούν, ίσως θα γίνουν αποδεκτά στο Μίνσκ την Τετάρτη, θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για κάποιες βιώσιμες πολιτικές εξέλιξεις. Ε, είναι κάτι πολύ πλοκό αυτό, δεν είναι εύκολο. Ξέρετε πόσο καιρό χρειαστήκαμε για να λυθεί το θέμα του κοσυφοπεδίου. Ε, χρειάστηκαν 10 χρόνια. Ας μην περιμένουμε λοιπόν γρήγορες λύσεις. Αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος, αν ξεκινήσει η πολιτική διαδικασία, αν πιστεύουμε ότι η θετική σκοπιά θα είναι ότι δεν θα έχουμε άλλους νεκρούς, νομίζω ότι ήδη αυτό είναι κάτι θετικό. Και αν χρειαστούν δύο-τρία χρόνια θα πρέπει να συνεχίσουμε. Όπως σε όλες τις κρίσεις τέτοιου τύπου. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι παρά τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση δεν θεωρούμε χθρό μας την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ε, και μερικές φορές αυτό λέγεται στον τύπο δεν είναι αλήθεια θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι και αυτή ανήκει στην ίδια ήπειρο με εμάς και ακούσαμε ότι στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει. Αυτό είπαν οι Βρυξέλλε. Όμω ακόμη και αν ισχύει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία. Ξεκολουθούμε να υπάρχουμε και θα είμαστε γείτονε στην ίδια Ήπειρο και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο τώρα εμείς να υπερβούμε την αμοιβαία ανταλλαγή κατηγοριών και να εξετάσουμε πώς μπορούμε να λύσουμε την κατάσταση αυτή, γιατί διαφορετικά αυτό θα μας οδηγήσει σε πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, βέβαια. Θα σας πρότεινα να έχουν 1,5 λεπτό οι συντονιστές και 1 λεπτό οι υπόλοιποι ομιλητές. Και έτσι μπορώ να κλείσω το κατάλογο ομιλητών. Κλείνω λοιπόν. Ο κύριος Πρέιντα έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Πρέντα. Χαίρομαι για την παρουσία σας σήμερα. δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν ο εισηγητής μας για τη Ρωσία να έρθει σε διάλογο μαζί σας στη χώρα σας. Ο κύριος Λαντσπέργης έπρεπε να πάει στη Μόσχα, αλλά δεν έχει γίνει δεκτός στο ρωσικό έδαφος. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται βίζα, επειδή έχει διπλωματικό διαβατήριο. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε εδώ. Κρίμα που δεν θέλετε να κάνετε μια συζήτηση σε ιδεολογικό επίπεδο, γιατί οι παρεμβάσεις σας τον Ιανουάριο ήταν καθαρά ιδεολογικές γιατί είπατε ότι η φιλελεύθερη ιδεολογία της δύση είναι μια μορφή ολοκληρωτισμού. Θα μπορούσα εκεί πέρα να κάνω μια πλήρη συζήτηση μαζί σας για να μπορέσω να καταλάβω λίγο καλύτερα τη θέση σας η οποία αναφερθεί και από τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Λαυρό προηγουμένως ε, πρόσφατα είπε ότι η Κρυμαία με τη δική της θέληση επανενσωματώθηκε στη Ρωσία, ότι δεν υπάρχουν ρωσικά στρατέματα στην Ουκρανία. Όλες αυτές οι δηλώσεις που τις γνωρίζουμε ήδη από την ε, δεκαετία του 50 και του 60, αυτός είναι ο ψυχρός πόλεμος κύριε Πούσκοφ, η συμπεριφορά σας. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που έχετε προέρχεται ακριβώς από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε σε πολιτικό επίπεδο τα προβλήματα αυτά δεν είμαστε στρατηγικοί εταίροι γιατί, γιατί το δικό σας καθεστώς είναι ένα καθεστώς το οποίο κινείται προς τη στρατικοποίηση. Θέλετε τον πόλεμο κύριε Πούσκοφ. Αν δεν θέλετε τον πόλεμο μπορείτε να το σταματήσετε εσείς. Δικιά σας ευθύνη δεν είναι η ευθύνη του Κιέβου, δεν είναι η ευθύνη της Ευρώπης. Αν θέλετε λοιπόν να σταματήσετε τον πόλεμο όπως είπατε, σταματήστε τον. Έχετε κάθε ευκαιρία να το κάνετε. Στις επόμενες ώρες, γιατί τα πράγματα είναι ήδη δύσκολα, Νομίζω θα έχετε τη δυνατότητα να δείξετε την καλή σας θέληση και να αποδεχτείτε μια πραγματική κατάπαυση του πυρός, η οποία θα οδηγήσει πράγματι στην κατάπαυση των εχθροπραξιών. Και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και κύριος Χάουιτ. Συμφωνώ καταρχήν απόλυτα με την ιδέα να προσκληθείτε εδώ όπως έπραξε ο κύριος Μπροκ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η πρωταρχική ανάγκη τώρα είναι να σταματήσουν οι μάχες. η απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης μπορεί να πάρει ένα κομβικό χαρακτήρα και νομίζω ότι ήδη έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και συμφώνησα με αυτά που είπε ο πρόεδρος μας στην παρουσίαση και την ενακτήρια, τις παρουσί... Ε, παρατηρήσεις τους. Αυτά που λέτε κύριε Πουσκόφ είναι διαφορετικά από αυτά που ακούμε από τον κύριο Λάφροφ και από τον κύριο Πούτιν και αυτά που βλέπουμε στη ρωσική τηλεόραση. Όταν βλέπουμε τι λέγεται εκεί για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι το ύφος το οποίο αναφέρατε είναι ακριβώς το ύφος που θα θέλαμε να έχουμε απέναντί μας αλλά δεν είναι το ύφος του διαλόγου λοιπόν, αλλά δεν είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μας αντιμετωπίζει η Μόσχα. Και ίσως θα μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί. Είπατε ότι είστε δεσμευμένου να βρείτε ειρηνικέ λύσεις. Αλλά αυτό δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τη χώρα σα δεν έχει σεβαστεί τι συμφωνίε. Αν θέλουμε πράγματι να έχουμε ειρηνική συμφωνία, θα πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην ακαιρεότητα. Και είναι πολύ σαφές για πολλούς από εμά ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη και ακαιρεότητα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση που θέλετε να δώσετε. Για μένα είναι παράξενο κύριε Πούσκοφ ότι μας ζητάτε να δεχτούμε μια λύση τύπου Κωσόβου όταν η κυβέρνηση της χώρας σας έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση για τη Σερβία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ τελειώνει ο χρόνο μου εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την πλευρά της συντηρητικής και μεταρρυθμιστικής ομάδας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Πούσκοφ ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και με τη δική μου χώρα βρίσκονται σε επίπεδο ψυχρού πολέμου σχεδόν αρχίζει στη χώρα μου μια ανάκριση για τον θάνατο του Λιβιτιένκο από ό,τι φαίνεται με διαταγές της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της ε, Ρωσίας. Εσείς έχετε τώρα μια ρεβανσιστική, αποχυσιστική για ορισμένε χώρες στρατηγική για να δημιουργήσετε νέα ρωσικά εδάφη και για μένα όλα αυτά είναι ένας πόλεμος επιθετικός εναντίον της ειρηνικής Ουκρανίας, ο Φίλιπ Κάμοντ, υπουργό εξωτερικών της χώρας μου, είπε ότι αυτό θυμίζει περισσότερο μια τυραννική ε, συμπεριφορά αυταρχικής κυβέρνηση και όχι μια δημοκρατική συμπεριφορά. Φυσικά εμείς θέλουμε μια δημοκρατική και ειρηνική λύση και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Μίνσκ τη ομάδα του Μίνσκ θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάτι τέτοιο, αλλά βλέπω ότι ο κύριο ε, Πούτιν και οι εκπρόσωποι του σε στρατιωτικό επίπεδο στο Ντονέτσκ και το Λουκάνσκ προτιμούν να δείξουν την υπεροχή της Ρωσίας σε επίπεδο στρατιωτικό. Πολλές από τι οβίδες που πέφτουν εκεί δεν έρχονται από τους αντάρτες όπως λέτε αλλά από τις ρωσικές πυροβολαρχίες. Η χώρα μου έχει υπογράψει τη συμφωνία της διαβεβαίωσης της, Βου... της Βουδαπέστης και δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Αν η χώρα σας τώρα ε, πάλι παραδιάσει μια συμφωνία στα πλαίσια της ομάδας του Μίνσκ και ζητά να υπάρχει ένας επίγειος διάδρομος ως την Κρυμαία ή το να κρατήσει τη Μαριούπολη ως σημαντικό λιμάνι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε τις ε, κυρώσεις και κυρίως να εμποδίσουμε κάθε πρόσβαση στις ρωσικές οικονομίες στη χώρα μου αλλά όπως λέει η Financial Times θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί στρατιωτική ικανότητα στην Ουκρανία να υπερασπίσει τον εαυτό σας. Διατηρείτε μια ψευδέστηση ότι υπάρχουν αντάρτες στην Ουκρανία. Κανένα δεν ξεγελάει αυτό. Και το γεγονός ότι εσείς έχετε ελάχιστη επιρροή απαραίτητος αυτό είναι αστείο. Θέλετε μια πανσλαβιστική Ρωσία, είναι κάτι που δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Εμείς δεν μπορούμε πια να έχουμε εταιρική σχέση με τη Ρωσία του Πούτιν. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πουσκόφ, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, 17 Απριλίου του 2014, ένα μήνα ακριβώς μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, δήλωνε τα εξή και παραθέτω. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Νόβα Ρωσία, ε, Λουγκάνσκ, ε, ε, Νικολάευ και Οδυσσός το επιτσάρου δεν ήταν ουκρανικά. Το επίκεντρο ε, ήταν Νοβοροσίσκ και η περιφέρεια ονομάζεται Νοβοροσία, Νέα Ρωσία. Εξ όσων ε, ε, κατανοώ και γνωρίζω είναι ένα τμήμα της ευρύτερης ρωσικής ειρήνης, Ρούσκι Κύριε Ρουσκόφ, που, που αρχίζει η, ε, ρωσική, ο ρωσικός κόσμος, το Ροσκιμίρ και πού τελειώνει και ποια είναι η σχέση σας με την πολιτοφυλακή που εσείς αποκαλείτε αντάρτες. Η Ρωσική Ομοσπονδία τους εφοπλίζει με το σύνολο του οπλισμού που χρησιμοποιούν για να ε, πολεμούν το Ουκρανικό κράτος. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν τέλει, μπορούμε να ακούσουμε και τι λέει κάποιο από τη Ρωσία στην Επιτροπή αυτή, γιατί μέχρι τώρα εγώ αυτά που έχω ακούσει μου προκαλούσαν φόβο να κάθομαι εδώ, γιατί οι συνάδελφοι εδώ στην Αφρική και στη ΣΕΤ ε, λένε ότι, ε, λένε ότι εσείς ε, στέλνετε τους στρατιώτες σας ε, να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ότι έχετε πολύ μεγάλους εξοπλισμούς και εν τέλει μπορώ να ακούσω και το λόγο της Ρωσίας ε, χωρίς να παρεμβαίνουν και να ερμηνεύουν στην αδελφή μου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είδαμε μια συνεχή αποσταθεροποίηση από την πλευρά της Ουκρανίας. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ε, σκόπιμη πρόθεση από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και από τον Ατλαντικό γειτονά. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια λύση προτείνετε εσείς, να μου την πείτε εσείς, όχι συνάδελφοι και κατόπιν η Ρωσία, ε, πώς θα έκρινε την παροχή όπλων ε, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτεών και αναφέρομαι σε κάποια όπλα που θα ήταν κατά τον τάξ ή φορητέ όπλα κατά των ε, αεροσκαφών. Εδώ παίρνουν τον λόγο όλοι κύριε Καούσο και ο Ρώσος πρέσβης όπως και άλλοι ε, της αντιπροσωπείας του κύριου Κάρας και μην δημιουργείτε την εντύπωση ότι για πρώτη φορά το τελευταίο δωδεκάμενο ακούμε τη φωνή της Ρωσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ναι, την, άποψή μου θα σας... Η κυρία Χάμς έχει τώρα το λόγο. Ναι, θα ήθελα κι εγώ να ε, σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχω να κάνουμε ερωτήσεις ε, ε, κάτι, με άμεσο τρόπο στον κύριο Πούσκοφ. Ε, ε, δεν μπόρεσα να πάω στη Μόσχα γιατί οι ρωσικές αρχές με εμπόδισαν να μεταβώ εκεί. Στο αεροδρόμιο του Σερεμέτιεβο με εμπόδισαν να ε, φτάσω στη Ρωσία δηλαδή. Και ακούγοντας αυτά που είπατε, ε, ε, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε και δεν η συμφωνία του Μίνσκ. Γιατί όλα αυτά που είπατε θα μπορούσαν να είναι πραγματικότητα βάσει της Συμφωνία του Μίνσκ. Επίσης, θέλω να γνωρίζω γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση ούτε αποφάσεις στη Ρωσική Δούμα για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Στην ομιλία σας αφήσατε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Ρωσία δεν ενέχεται καθόλου στη σύγκρουση εκεί. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ πολύ αμφιβάλλω, διότι όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται από τη Ρωσία. Για παράδειγμα, σήμερα ένας στρατηγικός γιατρός είπε ότι βεβαίως υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες που μάχονται στην Ουκρανία, είναι εθελοντές. Και όλο και περισσότερες φωτογραφίες βλέπουμε ε, να ε, υπάρχει εκεί ε, ρωσικό υλικό φορτηγά λοιπά. Η Δούμα, το Κρεμλίνο, πρόκειται να συμφωνήσει ε, με συμβιβασμό σαν αυτόν που επιτεύχθηκε πριν από μήνες το Μίνσκ. Και πόσο παραπέρα θέλετε να πάτε πέρα από τη συμφωνία του Μίνσκ ε, ως προς τα εδάφη και την επικράτεια. Γιατί θέλω να τονίσω τις πάρα πολύ σοβαρές ερωτήσεις που σας έκανα ο συνάδελφος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Πουσκόφ που παρευρέθηκε εδώ γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Συμφωνώ μαζί σας ε, όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί και δεν είναι άσπρο και μαύρο ε, ο πόλεμο αυτός ε, και ο Πλατώνας είχε πει ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Η ανάλυση σας ε, έλεγε ότι δεν είναι στρατιωτική λύση. Εγώ συμφωνώ, αλλά όχι μόνο το ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε και δεν θα έπρεπε αυτό να γίνει αποδεκτό ούτε από την ευρωπαϊκή πλευρά, ούτε οποιοδήποτε άλλο πρωταγωνίστη. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο μπραντεφέρ μιας μεγάλης υπερδύναμης ε, και μιας άλλη που θα ήθελε να γίνει υπερδύναμη και όλα όσοι και διακυβεύεται εδώ πάνε πολύ πιο πέρα από την κρίση στην Ουκρανία. Αλλά εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Υπό το φω αυτή τη κατάσταση, αν, αν υπάρχει μια πρόταση για να δοθεί μια μεγαλύτερη αυτονομία στι περιοχέ αυτέ, έχω παραδείγματο χάρη ε, κατά νου την περίπτωση του Τρεντίνο στη Βόρεια Ιταλία. Αν υπήρχε μια τέτοια πρόταση ε, τέτοιου είδου πέρα από το θέμα της Ομοσπονδίας, το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, πώς θα απαντούσε το Κρεμλίνο αυτή τη φορά θα υπήρχαν πραγματικές συνθήκες να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η παρουσία σας εδώ και η πρώτη μου ερώτηση είναι έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το πώς πρέπει να αξιολογήσουμε την πραγματικότητα που μας ανησυχεί όλους, θα πρέπει όλο το θέμα να αξιολογηθεί και σε σχέση με την αδυναμία των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, είναι αλήθεια ότι αυτή η πρωτοβουλία των δύο ηγετών της Γερμανίας και της Γαλλίας ε, κάποια στιγμή βγάζει εκτός παιχνιδιού ποιον θα έπρεπε να ε, ασκεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και και θα ήταν τα θετικά ενός ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεδομένου ότι η Ρωσία βάσει της ιστορίας και της γεωγραφίας είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μια μεγάλη αντίθεση, ένας μεγάλος ε, κίνδυνος εντός της Ευρώπης και πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι να λύνουμε τα ζητήματα μεταξύ μας ε, χωρίς να δεχόμαστε κάποιες επιρροές όποιον λέει ότι είναι έτοιμος να στείλει θανατηφόρα όπλα. Το δεύτερο θέμα, τηλεγραφικά, είναι αν θεωρείτε το εξής, ότι ε, πέρα από το θέμα της ακυριότητας ε, της κάθε χώρας με το οποίο συμφωνώ, ε, πρέπει να δούμε και το θέμα της αυτοδιάθεσης των λαών ε, και να φέρουμε και στην ρωσική μειονότητα στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Προτείνω ο επικεφαλής αντιπροσωπείας με τη Ρωσία και ο εισηγητής μας να μπορέσει να, λάβει το λόγο. Κύριος Λαντσβέργης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή που εστάλει να δει την επιτόπια κατάσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να μπει στην περιοχή. Κύριε Πούσκοφ, εσεί έρχεστε καλεσμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και παρουσιάστε τη δική σα θέση. Αυτό δείχνει και το χάσμα μεταξύ του δυτικού κόσμου και του δικού σα κόσμου. Είναι μεγαλύτερο το χάσμα γιατί η Ρωσία δεν σέβεται τι υποχρεώσει που έχει ίδια προσυπογράψει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1.435 αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν εφαρμόζει η Ρωσία αμέσως μετά από την είσοδό της στον ΠΟΕ η Ρωσία έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις της για το ελεύθερο εμπόριο και είναι σε σύγκρουση για πολλά θέματα με την Ευρώπη. Το μνημόνιο της ε, Βουδαπέστης, ε, η απόφαση τελική του, της πράξης του Ελσίνσκι, χάρτης του, των Ηνωμένων Εθνών, πάρα πολλές πράξεις που έχει υπογράψει η Ρωσία δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι <clears throat> η Ρωσία δεν έχει κινήσει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι για να εφαρμόσει την συμφωνία του Μίνσκ. Πώς μπορείτε να φανταστείτε οποιαδήποτε σχέση με τη λύση όταν απορρίπτετε την καλή μας ε, θέληση, κάνετε συμφωνίες που δεν τις δέχεστε και απορρίπτετε το κράτος δικαίου και την δημοκρατική διαδικασία. Ο επόμενος ομιλητής. Ένα λεπτό λοιπόν οι υπόλοιποι ομιλητές. Ο κύριος Πίκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πούσκοφ για τα σχόλιά σας. Είπατε ότι στην αρχή κάθε σύγκρουσης ξεκινούν, ξεκινάμε μικρά πράγματα και μετά αρχίζει και κλιμακώνεται. Σα ότι το πυρηνικό πλωστάσιο τη Ουκρανίας πήγε στη Ρωσία με αντιστάθμισμα μια συμφωνία που πρέπει να εξασφαλίσει το σεβασμό των, ε, της εδαφικής της ε, Ουκρανίας. Θεωρείτε ότι δεσμεύεται η Ρωσία, είναι το ερώτημα μου, από το μνημόνιο της Βουδαπές του 1944, κυρία Καλνιέτα. Κύριε Πουσκόφ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα ακυρώσει η Ρωσία το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή μήπω προτιμάτε να μην το κάνετε γιατί φοβόσαστε ότι θα έρθει κάποια μέρα όπου οι Ρώσοι στρατιώτες, η ελίτ των Ρώσων στρατιωτών που πολεμάει στην Ουκρανία θα είναι ενώπιον του δικαστηρίου λόγω των εγκλημάτων τους εκεί. Ο κ. Φλέκενστίν. Κύριε Πουσκόφ, είπατε ότι η στρατηγική εταιρική σχέση σα ε, ε, ε, σας είπαν ότι καταργήθηκε. Ε, νομίζω ότι αυτό μας λείπει περισσότερο από όσο πιστεύετε, γιατί θα ήταν απαραίτητος ε, ε, επεγόντως κιόλας απαραίτητο να υπάρχει τέτοια συμφωνία για να μπορούμε να λύνουμε ό,τι θέματα έχουμε μεταξύ μας. Είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό γρήγορα. Συμφωνώ και εγώ το ίδιο πιστεύω. Αλλά δεν θέλουμε να παραβλέπουμε και να παρακάμπτουμε την επόμενη παγωμένη σύραξη. Υπάρχει μια προϋπόθεση για να ε, τα λύσουμε πολλά ε, από τα θέματα που μας ενοχλούν με αμοιβαιότητα. Είπατε ότι είστε υπέρ της εκεχηρίας και εγώ. Επιτρέψτε μου και να με συμπαθάτε που είμαι ε, επιφυλακτικός και σας παρακαλώ να μην μας απογοητεύσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πουσκόφ. καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ για το διάλογο που έχετε μαζί μας. Για να συνοψίσω τα όσα είπατε, δύο προτάσεις. Λέτε ότι έχει έρθει η ώρα για κάτι καινούριο και ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά και σας ερωτώ. γιατί ε, ε, εισαγάγατε εσείς τον πόλεμο εκεί. Είναι εισαγόμενος πόλεμος, υβριδικός στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία ανέκαθεν ε, διέψευδε τη συμμετοχή της. Αλλά ποτέ δεν έβλαβα απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία ότι πού τα βρήκανε αυτά τόσο βαρέο πλισμό και όλο αυτό το υλικό που έχουν οπλισμο και ολο αυτο το στρατιωτικό. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Και δεύτερη ερώτηση πότε θα απελευθερωθεί η Νάτια Σευτσένκα που είναι μέλος ε, της Ουκρανικής ε, Βουλής και του Συμβουλίου της Ευρώπης που με κάτι θολές κατηγορίες την ε, έχουν κρατούμενη στη Μόσχα παραβιάζοντας κάθε διεθνή κανόνα. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Εγώ πιστεύω ότι είναι τεράστιο λάθος να κρίνουμε τη Ρωσία, να τη βάζουμε σε δίκη, όπως κάνουν ορισμένοι από εμάς, πρέπει να βρούμε μια πολιτική λύση σε ένα πρόβλημα στρατηγικά τεράστια σημασία. Ε, δεν ξέρω και ήμουν ανταποκριτής για 30 χρόνια. Έκανα ε, ένα πόλεμο που να κάνει κάποιος ε, από υποχρέωση σε τρίτους. Υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι στην Ανατολική Ουκρανία και σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό. είδαμε το 52% του ποσοστού πήρε και όταν ο Υπουργός όταν ε, ο Υπουργό Άμυνα τη Ουκρανία ε, καλεί να πάρουν τα όπλα, ε, μόνο το 20% ανταποκρίνεται. Εδώ πρέπει να βρούμε ένα τρόπο αποκλιμάκωση. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Καταρχήν, η Ρωσία ε, θεωρεί ότι ξεκολουθεί να έχει το πρωτόκολλο τη Βουδαπέστη. Ε, σημαντικό ζήτημα. Δεύτερον, ποια λύση έχετε κάτω νου για τον Τόνμπα και για την Κρυμαία. Και συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να υπογράψετε τη συνθήκη ε, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όμως εγώ θα ήθελα αυτό να το ζητήσετε και για το Ισραήλ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πούσκοφ σίγουρα μας χωρίζει τεράστια ιδεολογική απόσταση ίσως ε, μεγαλύτερη από αυτή που με χωρίζει με τον κύριο Μπρόκ και με άλλους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής. Εγώ θέλω να επενέσω το θετικό του ύφου σα και το γεγονός ότι είπατε κάτι πάρα πολύ λογικό, ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Μακάρι ορισμένα από τους συναδέλφους που να μιλούσαν με τον ίδιο τρόπο σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι το εμπριστικό ύφο μπορεί να είναι καλό σε μια συνέλευση φοιτητών φοιτητών αλλά όχι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ το ξέρουμε όλοι, ακόμα και αν μην το αναγνωρίσουμε, ότι οι διεθνεί σχέσει βασίζονται περισσότερο στη γεωπολιτική παρά στην ιδεολογία ή στη φύση ή στι συμπάθειε για ένα πολιτικό καθεστώ. Και έχουμε την ανάδυση σε γεωπολιτικό επίπεδο τη Ρωσία ω νέα δύναμη που είναι κάτι που είναι γεγονό. Υπάρχουν κάποιε πολιτικέ δυνάμει οι οποίε θέλουν να ανακτήσουν μια διαφορετική Ευρώπη και θέλουμε να έχουμε μια βασική σχέση σεβασμού, συνεργασίας αλλά και σεβασμού, με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου με τη χώρα σας. Είναι ακριβώς οι σχέσεις που θέλουμε να έχουμε και όχι αυτές που έχουμε με τις ΗΠΑ που δεν διέπονται πάντα από το σεβασμό της ε, διεθνούς νομιμότητας. Thank you, Mr. Rishkov, Ευχαριστώ κύριε Ρουσκόφ ήρθατε στο κοινοβούλιο. Sorry, misspoke. Mr. thank Σας ευχαριστώ, έλεγα κύριε Πουσκόφ. Θέλω να σας ρωτήσω. Θα εργαστείτε ε, χωρίς ε, καμία ε, επιφύλαξη για κατάπαυστα για να μπορούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ταξιδεύουν στη Ρωσία και στη Μόσχα. Επίσης, θα βεβαιωθείτε ότι η συμπεριφορά σας ευθυγραμμίζεται πλήρως με ε, το χάρτη των Παρισίων. Και όταν ο Σέρβος ε, επικεφαλής του ΟΑΣΕ ε, επέκρινε τους λεγόμενους αντάρτες γιατί δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε εκεχηρία με βάση τη συμφωνία του Μίνσκ. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε. Hvala lijepa predsjedavajući kolega Brok, e, gospodine Puškov, hvala što... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπροκ. Κύριε Πουσκόφ, σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε σε αυτή την επιτροπή σήμερα. Θέλουμε να σας ε, ρωτήσουμε πιστεύετε ότι οποιαδήποτε όμορφη χώρα της Ρωσίας ε, που επιλέξει τον Ευρωπαϊκή Οδό θα αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο σενάριο. Ποια είναι η θέση της Ρωσίας σε ό,τι αφορά ε, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και πιστεύετε ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας ε, πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζεται στη Ρωσική Δούμα όταν ε, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Επίσης, ε, μας υπενθυμίσατε τι συνέβη με το Μιλόσεβιτς τη δεκαετία του 90. Μια τέτοια κατάσταση φυσικά δεν είναι καλή για μια επίρροπη που θα συνεχίσουμε να ζούμε όλοι μαζί στο μέλλον. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε με κάθε σεβασμό προς τον καλεσμένο. Θα ήθελα να μιλήσω ρωσικά γιατί υπάρχει μετάφραση. Εγώ εκπροσωπώ τη Λετωνία και η χώρα μου. Ίσως είναι αυτή που ξέρει καλύτερα πώς το πάγωμα των σχέσεων με τη Ρωσία έχει άμεσες επιπτώσεις στη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εχθρός σας, το ξέρετε αυτό. Αλλά πέστε μου ποια είναι τα βήματα που είναι έτοιμη να κάνει η Ρωσία για να μπορέσουμε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αν υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ καταρχήν. Σας ευχαριστώ που δεν προσπαθήσατε να μας πείσετε ότι ο στρατός σας και το σας δεν είναι στην Ουκρανία. Δεύτερον, όπως και άλλοι συναδελφοί, ε, το να ε, απελευθερώσετε την αντίστοιχα αμέσω δεν έχετε δικαίωμα να την κρατάτε γιατί η Ρωσία δεν έχει επιτρέψει πρόσβαση ε, του ΑΣΕ στην ε, περιοχή και γιατί δεν είχε επιτρέψει ε, τα ντρόν ε, να πάνε εκεί για να δούμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Η επόμενη ερώτηση αναφερθήκατε στην εθνοτική σύνθεση του Λουκάνσκ και του Ντονέσκ με το ίδιο ε, επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για το Κίεβο ή και για άλλες περιοχές. Ε, δηλαδή, αν χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο επιχείρημα, πού ακριβώς θα σταματήσετε, ποιες ε, εγγύσεις μπορείτε να μας δώσετε και διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθεί κάπου, θα έχει και ένα τέλος η όρεξή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μελανσό. Κύριε, ο πρόεδρος Μελανσό, ναι. Σας ευχαριστώ κύριε, αγαπητέ κύριε πρόεδρε. Με όλο το σεβασμό που έχω για σας, κύριε πρόεδρε, δυστυχώς δεν σύμφωνο με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Πούσκοφ που είναι παρόν εδώ. Δεν θα πρέπει να πιστέψει ότι όλη η ευρωπαϊκή ε, κοινή γνώμη έχει την ίδια άποψη με αυτά που ακούσατε εδώ. Εδώ, στη Γαλλία, όλη η κοινή γνώμη μέχρι και ο Πρωθυπουργό μα, τόνισαν δεν χρειάζεται ιστερία κατά της Ρωσία. κάνε δεν θα κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας παρά μόνο κάποιος τρελός και δεν θα επενέβαινε κατά στην Ουκρανία να επιτεθεί σε ποινικού σταθμού όπως είπαν ορισμένοι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ε, επεμβάσεις. Κανείς δεν λέει τίποτα για την επέμβαση των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απόλυση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όλα αυτά τέλος πάντων είναι απλώς μια ευχάριστη φλιαρία. Το Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ των προέδρων μας, των προέδρων τη δική μου Χώρα και τη δική σα. Θα ήθελα να ξέρω τι θα κάνει το δικό σα κοινοβούλιο στη συμφωνία η οποία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αυτό το Σαββατοκύριακο θα υλοποιηθεί από με μία απόφαση και η Ρωσία θα εξασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και θέλω να σας πω ότι οι, οι συμπατριώτες μου είναι πάντα ευγνώμονες για το ρόλο που έπαιξε η Ρωσία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ε, απελευθέρωση της χώρας μας και κάνει δεν πρέπει να ξεχάσει τους 20, τα 20 εκατομμύρια νεκρών της Ρωσίας στην υπηρεσία της ελευθερίας. Mr. Mélenchon, Κύριε Μελανσόν, για την απελευθέρωση της Γαλλίας, ξέρει, ήταν και κάτι Άγγλοι και κάτι Αμερικανοί εκεί, τους οποίους μόλις επιτεθήκατε. Και παρακαλώ να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Στην Ορμανδία, έτσι, στην απόβαση ήταν κάτι Άγγλοι και κάτι Αμερικανοί. Δεν τους ξεχνώ κύριε Πρόεδρε, αλλά ε, ε, δεν θα πρέπει να ξεχάσετε κι εσείς ε, τους Ρώσους. Stop θα, πρέπει να σας πω κύριε ότι αν επρέσβευα τα ίδια με εσάς εγώ θα, θα αμφέβαλα και θα αναρωτιόμουν αν είναι λανθασμένη ή όχι η απόψη μου. Ο συνάδελφος Σοπράτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ε, με έχει οδηγήσει σε ευθυμία αυτό που ακούω από κάποιους συναδέλφους που δίνουν μαθήματα στη Ρωσία ελεύθερης κυκλοφορίας ε, όταν Υπάρχουν ε, και λίστες για κυρώσεις για πολλούς Ρώσους πολίτες. Αρκετά εύθυμα είναι αυτά που ακούμε εδώ μέσα. Ε, μας αρέσει πολύ να δίνουμε μαθήματα χωρίς να εφαρμόζουμε όμως τις ίδιες μας τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές. Ένα αυτό. Δεύτερο, να θυμίσω λίγο κάτι από την ιστορία του 1981. 1981 Γαλλία και Γερμανία θέλησαν να φτιάξουν αγωγό φυσικού αερίου προς τη Σιβηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις. Η Γαλλία η Γερμανία ενώ ήταν ε, τότε ψυχρός πόλεμος αντιστάθηκαν και το 1982 αναγκάστηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε να υποκληθούν και να άρουν τις κυρώσεις. Και ήταν ψυχρός πόλεμος. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λιγότερη εξάρτηση από την ΕΟΚ τότε, από τους Αμερικανούς. Και παρακαλώ συνάδελφοι να σκεφτούμε για ποιο λόγο σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση... Τέλειωσε ο χρόνος σας λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ σταματήστε. Ε, η απάντηση είναι στην επιθετικότητα του κυρίου Πρέντα. Είναι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η απάντηση. Ένα λεπτό έκαστος είπαμε. Εδώ η διαφορά. Εδώ στο κοινοβούλιο μπορεί οι πάντες να ομιλούν. Και ε, ακούσαμε πολλούς ε, ομιλητές που δεν είναι στην πλειοψηφία του ψηφίσματο. Γι' αυτό είμαστε ελεύθερο κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να το εκτιμάτε ότι όλοι μιλάτε. Κυρία Γκόμε. Καλώ ήρθατε, κύριε Πουσκόφ. Θέλω να σα ρωτήσω γιατί δεν δέχεται η Ρωσία ότι είναι μέρο σε αυτόν τον πόλεμο και αναγνωριστείτε ότι το Ντόνμπας είναι μέρο τη Ουκρανία. Αυτό ισχύει και για τη Μαριούπολη. Θα ήθελα να μου πείτε και για την Κρυμαία ρωτήθηκε το θέμα αυτό και είπατε ότι χρειάζεστε εγγύησεις γιατί να, να λειτουργήσει η συμφωνία του Μίνσκ. Ποιες εγγύησεις χρειάζεστε. Κύριος Χαζηγεωργίου παρακαλώ. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Πουσκόφ εδώ. Μικρόφωνο, μικρόφωνο κύριε Χαζηγεωργίου. Εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ από το ψυχροπολεμικό κλίμα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη ως να μην έχουμε πάρει ποτέ μαθήματα από τους πολέμους και τα εκατομμύρια των νεκρών. Απόδειξη δε αυτού του ψυχροπολεμικού κλίματος ήταν και κάποιες στιγμές μέσα σε αυτή την ίδια την αίθουσα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις έφεραν οποιοδήποτε αποτέλεσμα και πολύ περισσότερο διαφωνούμε με την αποστολή νέων όπλων από τις ΗΠΑ ή από το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτό θα φέρει περισσότερο αίμα και τίποτε άλλο στην ε, περιοχή αυτή. Η αναφορά στο Βιετνάμ νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή αναφορά εκ μέρους του κυρίου Μπουσκόφ αλίμονο αν δούμε ένα Βιετνάμ μέσα στις τάξεις, ε, της, μέσα στον χώρο της Ευρώπης. Κλείνω με δύο ερωτήσεις. Ποιες επιπτώσεις έφεραν οι κυρώσεις στην ε, Ρωσία, κύριε ε, Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών και επειδή αναφερθήκατε σε Ομοσπονδία θέλω να μου πείτε αν εννοείται και την Κρυμαία. Ο κ. ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ κύριε Πούσκοφ. Πάντα πιστέψαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις εδώ του 21ου αιώνα που είναι η τρομοκρατία, η ακεροφροσύνη κτλ. Τα θέματα της ενέργειας, της οικονομίας, της κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς, για να μπορούμε να έχουμε συνεργασία χρειάζονται και οι δύο πλευρές να συνενούν. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ρωσία θα παραμείνει πιστή στις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει. Τρία ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα. Πιστεύει η Ρωσία ότι θα πρέπει να τηρήσει το μνημόνιο του, της Βουδαπέστης του 1994. Πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια συμφωνία μεταξύ του πρεσβυτέρου κ. Μπούς και του κ. Γκορμπατσόφ σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη που θα πρέπει να γίνουν δεκτά ή όχι στον ΝΑΤΟ. Γιατί ορισμένοι λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του από αυτή την άποψη. Και τρίτον, δεν συμφωνείτε ότι υπάρχουν πολλές ακροδεξίες και ακροαριστερές δυνάμεις σήμερα στην Ευρώπη. Κύριε Πούσκοφ. Τα λεπτά λέει ο πρόεδρος. Alors voilà, j'ai 7 minutes. Έχω 7 λεπτά για να απαντήσω σε όλους αυτούς τους ομιλητές, δε κύριος Ρίσκο. Euh, Θα σταθώ στα πιο σημαντικά στοιχεία. Θα απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, όχι βέβαια σε όλα τα ερωτήματα, γιατί σε 7 λεπτά πραγματικά δεν προφθαίνω. Ναι. Ο πρόεδρος μου είπε 7 λεπτά. Ξεκινώ με το ερώτημα του πότε η Ρωσία θα ακυρώσει την προσχώρησή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. <clears throat> Ίσως όταν το κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως όταν το κάνει και η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία δεν έχει κυρώσει αυτή την συμμετοχή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπάρχουν πολλές χώρες, δεν είναι μόνη η Ρωσία και δεν πρέπει να δακτυλοδεικτείτε. Επίσης, υπήρξε μια δήλωση ότι οι βομβαρδισμοί έρχονται κυρίως από, τα, από τη ρωσική πλευρά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι βομβαρδισμοί γίνονται κυρίως από τον Ουκρανικό στρατό. Το πρόβλημα είναι ότι αν υπήρχε βομβαρδισμός μόνο στρατιωτικών θέσεων των ε, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι πόλεμος, αλλά βομβαρδίζονται πόλεις ολόκληρες. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν 7-8 νεκροί στον Τονέσκ Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι αυτές οι, αυτοί οι βομβαρδισμοί, αυτές οι οβίδες έρχονται από την Ουκρανική πλευρά. Σας Λέω ότι αυτό είπε η Human Rights Watch που είναι ένας φορέας ο οποίος κατά την άποψή μου είναι αρκετά αμερόληπτος και έχει κατηγορήσει τον Ουκρανικό στρατό για χρήση βομβών διασποράς. Τρεις φορές. Το έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά τα ευρωπαϊκά ε, όργανα, τη χρήση όπλων που είναι απόλυτα παράνομα. Παρ' όλα αυτά τα χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα οι Ουκρανοί. Ακόμα και βαλιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν από τον στρατό τη Ουκρανία. Αυτό το έχει αναγνωρίσει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτά είναι γεγονότα. Όταν σα λέω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μπορούν να νομίζουν ορισμένοι. Είναι πράγματα που πρέπει να τα λάβετε υπόψη. Για την Κρυμαία επίση. Το θέμα τη Κρυμαία επανέρχεται πάντα. Πρέπει να σα πω για μια ακόμα φορά. Δεν πρόκειται να αναφέρω τι ρωσικέ πλευρέ γιατί υπάρχουν και άλλε πηγέ έγινε από το πρακτορείο Γκάλοπ μια δημοσκόπηση τον Απρίλιο 83% αυτών που απάντησαν σε αυτή τη δημοσκόπηση είπανε ότι το δημοψήφισμα στην Κρυμαία αντανακλούσε τις απόψεις των κατοίκων της Κρυμαίας. Στις 8 ε, Μαΐου το Q Research Center, πάλι αμερικανικός φορέας, 91% των απαντώντων είπαν ότι το δημοψήφισμα ήταν αμερόληπτο και ελεύθερο. Αν έχετε λοιπόν ερωτήματα, μιλήστε στην Q Research, μπορείτε να τους ε, καλέσετε να σας εξηγήσουν. Πριν από τρεις εβδομάδες, μια γερμανική ομάδα δημοσκοπήσεων έκανε μελέτες για την Κρυμαία και έδειξαν ότι 93% των κατοίκων της Κρυμαίας υποστηρίζουν την ενοποίηση της Κρυμαίας με τη Ρωσία. <clears throat> Αυτά όμως έρχονται από δημοσκοπικούς οργανισμούς της Δύσης. Δεν τα έχουμε εφεύρει εμείς. Επομένως όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει. Είναι γεγονός αυτό. Δεν μπορείτε να το παραγνωρίσετε. Πρέπει να το δείτε κατάματα. Είναι δικό σας πρόβλημα. Όταν κοιτάζει κανείς τον καθρέφτη, βλέπει κάτι πρέπει να το λάβει υπόψη σοβαρά. Παρακαλώ, λέω ο πρόεδρος. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα. Κατά πόσο οι χώρες που είναι γειτονικές της Ρωσίας θα πρέπει να νιώθουν φόβο για τη, Ρωσία, για τη Ρωσία, για ρωσική ισχύ. Κατά τη δική μου άποψη δεν υπάρχει καμία απειλή για τις όμορες χώρες της Ρωσίας. Καμία. Καμία απειλή. Το ξαναλέω, καμία απειλή δεν υπάρχει. Η Αρμενία. Μα εδώ είσαστε παράλογος. Είναι απόλυτα παράλογο αυτό που λέτε. Αν μελετήσετε λιγάκι το θέμα και ελάτε μετά στη Μόσχα να τα ξαναπούμε. Όχι, θα σας δώσουμε. πάτε με τηλέφωνο και θα κανονίσω να έχετε βίζα. Η Ρωσία δεν είναι κίνδυνος για την Ευρώπη, ούτε για τη Δύση ο κίνδυνος είναι αλλού. Ο κίνδυνος έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Είναι το Ισλαμικό κράτος. Αυτό αποκεφαλίζει τους δυτικούς δημοσιογράφους. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά η Ρωσία. Κάτι ακόμα θέλω να σας πω. Υπάρχει προπαγάνδα <clears throat> όταν ο κύριος Ομπάμα και ορισμένοι βουλευτές ε, συγκρίνουν με το Ισλαμικό Κράτο στη Ρωσία καθώς και με τον ιό έμπολα. Αυτό είναι σκανδαλώδε. Αν δείτε τα πράγματα κατάματα, θα, καταλαβα... θα καταλάβετε τη Ρωσία η οποία ήταν η πρώτη που έδωσε τη βοήθειά τη στις Ηνωμένε Πολιτείε μετά από την τραγωδία τη 11 Σεπτεμβρίου 2001. Το ξέρουν αυτό οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και ο George Μπού ιό το θυμάται πολύ καλά. Μετά από αυτά που έγιναν επίση στο Παρίσι, Πρόσφατα, τα γεγονότα του Σαλί έχουμε και εκεί πάλι εκφράσει τη, θέλησή μας να αγωνιστούμε μαζί με την Ευρώπη κατά της τρομοκρατίας. Ήταν δηλώσεις του Πούτιν και του Λαυρόφ. Αν ζητήσετε από τις ειδικέ σας, από τις υπηρεσίες σας πληροφοριών, θα δείτε ότι πάντα υπήρχαν ανταλλαγές πληροφοριών και συνεργασίες και η Ρωσία πάντα πληροφόρησε τις δυτικές υπηρεσίες για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες στη Δύση. Και ξέρω τι λέω εδώ. Για τις σχέσεις με την ΟΑΣΕ. Πιστεύουμε ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την ΟΑΣΕ. Πάντα υπήρχαν βέβαια προβλήματα, πάντα υπάρχουν προβλήματα η ΟΑΣΕ. Θα είναι παρούσα στη Ρωσία την επόμενη εβδομάδα η επικεφαλής της κοινοβουλευτική συνέλευση τη ΟΑΣΕ θα είναι την Πέμπτη στη Ρωσία αφού, πέρασε από το, αφού πέρασε από το Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω θα μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί της και εξάλλου στο Μίνσκ θα υπάρξει η υπογραφή ενό εγγράφου από του αρχηγού των κρατών μα. Η κυρία που είπε ότι δεν ε, μπόρεσε να μπει στη Ρωσία. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι. Δεν αρχίσαμε εμείς να βάζουμε του βουλευτέ σε μαύρε λίστες. Αυτό δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Ναι, για το Μίνσκ. Η συμφωνία του Μίνσκ δεν φτάνει. Λέτε ότι παραβιάστηκε, μα έχει παραβιαστεί ήδη πολλές φορές και από τι δύο πλευρές. Γι' αυτό δεν φτάνει η συμφωνία του Μίνσκ. Χρειαζόμαστε κάτι πιο σταθερό που να βασίζεται σε αυτή τη συμφωνία και όταν μιλάτε για τη συμφωνία του Μίνσκ ξέρετε ότι το αεροδρόμιο του Ντονέσκ για το οποίο πολεμούσε ο Ουκρανικός στρατός μέχρι πρόσφατα έπρεπε να είχε απελευθερωθεί και εκενωθεί το Σεπτέμβριο. Γιατί αυτό ήταν μέσα στι συμφωνίε του Μίνσκ. Δεν θέλω να μπω λοιπόν σε διαμάχη για κάθε συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Όταν μιλάμε όμω για τι συμφωνίε του Μίνσκ σαν βίβλο, θα πρέπει καταρχήν να τι ξέρουμε καλά αυτέ τι συμφωνίε και δεύτερον θα πρέπει να δούμε ότι παραβιάστηκαν και από τι δύο πλευρέ. Γι' αυτό χρειάζεται μια διεθνή παρέμβαση γιατί όσοι έχουν τα πράγματα τώρα επί τη βάση των συμφωνίων του Μίνσκ δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και τέλος. Το μνημόνιο τη Βουδαπέστης τώρα. Ερχόμαστε στην ουσία τώρα του προβλήματος. Η ουσία είναι, είναι το θέμα του διεθνούς δικαίου, κατά την άποψή μου. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο. Όταν το Κωσυφοπαίδιο αποχωρήθηκε από τη Σερβία, όπως ξέρετε το Βελιγράδι δεν έδωσε την έγκρισή του. Έγινε κάτι ενάντια στη θέληση του κράτους το οποίο συμπεριλαμβάνεται το Κόσοβο και είναι και πόλεμος εναντίον της Σερβίας. Αυτό ήταν παραδίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι φανερό. Η παραδίαση λοιπόν του διεθνούς δικαίου επίσης ήταν και η εισβολή στο Ιράκ. 27 χώρες ευρωπαϊκής της Ευρώπης ήταν κομμάτι αυτής της ε, επιχείρησης, είτε με στρατεύματα είτε με υποστήριξη. Και αυτό ήταν παραδίαση του ανθρωπίνου δικαίου. Όλοι το ξέρουν τώρα. αυτό που θέλω να πω. Και η Λιβύη επίσης, ξέρετε ότι υπάρχει και άλλη αντιμετώπιση για το ψήφισμα 1973 για τη Λιβύη. Δεν έδινε το δικαίωμα βομβαρδισμού της Τριπολίτιδος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε μια μεγάλη κρίση για το διεθνές δίκαιο. Και αν υπάρχουν χώρες οι οποίες παραβιάσουν το ανθρώπινο το διεθνές δίκαιο, δεν μπορούν να περιμένουν από τους άλλους να μην κάνουν το ίδιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαλέξουμε και να πούμε αυτό το ψήφισμα ή το, το τάδε μνημόνιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τα άλλα δεν είναι. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Πούσκοφ. Δεν μπορούμε να πούμε <clears throat> ότι εδώ λειτουργεί το διεθνές δίκαιο και αλλού δεν, δεν λειτουργεί. Επειδή μας αρέσει μια περίπτωση και όχι στην άλλη. Αυτά που σας λέω λοιπόν δεν σας τα λέω αυτό θέλω να σας πω ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό μάτι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σειρά κανόνων που θα μας επιτρέψουν να ξέρουμε πού βρισκόμαστε γιατί αν οι κανόνες παραβιάζονται από τους μεν δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους δε να τους σέβονται. Όταν έγιναν τα γεγονότα του Κωσόβου η Ρωσία είπε άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και μου λέει ο Έλμαρ Μπρόκμα είναι ειδική περίπτωση, μα υπάρχουν πάρα πολλές ειδικέ περιπτώσεις τότε. Και η κρυμμένη είναι ειδική περίπτωση. Θα υπάρξουν και άλλες ειδικέ περιπτώσεις. Αν δημιουργείται ένα προηγούμενο λοιπόν, θα πρέπει να περιμένετε ότι θα υπάρξουν και άλλες ειδικέ περιπτώσεις. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, θέλω να προσκαλέσω μια ομάδα βουλευτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κλείνει πάλι το μικρόφωνο του ομιλητή. Θα ήθελα να έρθει μια ομάδα βουλευτών στη Μόσχα για συζητήσεις για τα προβλήματα αυτά. Είχαμε την πρακτική να έχουμε ανταλλαγή αντιπροσωπιών. Το Μάτιο πέρσι είχαμε, ναι, στο Στρασβούργο και είχαμε κάνει συζητήσει εδώ. Τώρα είναι δική σα σειρά να έρθετε στη Ρωσία και θα χαρούμε πάρα πολύ να σα δεχτούμε στη Ρωσία Πεςτε μου πότε θα θέλετε να έρθετε και θα εξασφαλίσω βίζα για όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου μια στιγμή μην φύγετε. Κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, είναι γεγονός ότι ε, η Ρωσία έχει εργαστεί και συνεργαστεί επικοδομητικά σε πολλά θέματα. Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, οικονομικά ζητήματα, εμπορικά και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράκ τη Συρία και το Ισλαμικό κράτος και τα λοιπά και άλλα τεινά. Αυτό δείχνει πολύ περισσότερο ότι έχει σημασία να έχουμε καλές σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Και αυτό γίνεται μόνο με το σεβασμό του ε, διεθνούς δικαίου. Έχει όμως μια τεράστια διαφορά Κωσυφοπαίδιο και ε, Κρυμαία. Επιτέθηκε στο Κωσυφοπαίδιο ε, η Σερβία και έκανε γενοκτονία ενώ άλλη είναι η Κρυμαία και ο ρωσικός πληθυσμός εκεί. Υπάρχει μια δραματική διαφορά και παρακαλώ να μην γίνονται συγχύσεις. Ε, δεν μπορούμε, δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα πράγματα. Και επίσης δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να ε, δικαιολογεί την παραβίαση της εδαφικής ακαιρεότητας μιας χώρας. Δεν έκανε τίποτα η Ουκρανία που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε. Βάσει όλων αυτών θα πρέπει να συζητήσουμε οπωσδήποτε. Επιστεύω ότι είναι αποφασιστική ε, η συγκυρία για να βρεθεί ένα αποτέλεσμα την Δετάρτη. Θα πρέπει να δεχτεί και η Ρωσία ότι είναι ενεχόμενο μέρος ε, ε, ε, εμπλέκεται εκεί, έχει προσαρτήσει έδαφος, έχει στρατεύματα που πολεμούν και θα πρέπει να συνεισφέρει γιατί είναι εμπόλεμη πλευρά. Θα πρέπει να το αναγνωρίσει η Ρωσία ότι είναι ένα ενεχόμενο μέρος και αυτό είναι κλειδί. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της ότι μα δεν ε, συμμετέχουμε εμείς εκεί στις εχθροπραξίες. Είστε εμπόλεμο ε, μέρος. Και θα πρέπει βεβαίως να ε, συνεργαστείτε για να λυθεί αυτή η σύγκρουση. Χαίρομαι που έγινε σήμερα αυτή η συζήτηση και ελπίζω να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Αλλά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφής. Στην ευρωπαϊκή τάξη σιρήνης ε, ανήκει η αναγνώριση και η υλοποίηση και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Πέρε.